Κυρίες και κύριοι, ψηφοφορίες. Καθίστε παρακαλώ, διότι αρχίζουν, όσον ούπο. Θα ψηφίσουμε τώρα, σύμφωνα με την απλουστευμένη διαδικασία, την έκθεση κυρίας Κιούστιγκερ. Ε, εθελοντική Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας. Το λόγο έχει η συγγήτρια, ε, κυρία Κιούστιγκερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Στις δύο πρώτες ψηφοφορίες έχουμε δύο εθελοντικές συμφωνίες ε, της Ένωσης με τη Λιβερία Φενός και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία Αφετέρου οι συμφωνίες ε, αποσκοπούν ε, σε ένα σύστημα πιστοποίησης για να βλέπουμε ότι η ξυλία αυτή θα είναι αντικείμενο νόμιμης ε, υλοτόμησης και νόμιμης εμπορίας. Είναι πολύ σημαντικός κλάδος της οικονομίας στην Αφρική το ξύλο και δίνεται η ασφάλεια στις ευρωπαϊκές εταιρείες και στους ευρωπαίους καταναλωτές ότι είναι νόμιμη η ξυλία αυτή και η εμπορία της. Ευχαριστώ. Ε, στους τους που συνεισέφεραν ε, τα μάλα για την προστασία του περιβάλλοντος, την αηφορία και την συμπερίληψη όλων των ομάδων του πληθυσμού σε αυτές τις χώρες που έχουν ε, πληγεί πάρα πολύ και από εμφυλίες σειράξεις. Ωραία, λέει ο πρόεδρος και περνούμε στην ψηφοφορία. Ψήφι υπέρ της έκθεσης και ο κατά αποχές εγκρίνεται. Η επόμενη έκθεση της κυρίας Κένστιγκερ, το ίδιο θέμα, αφορά τη Συμφωνία τελικής Σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Λιβερίας. Ψήφιπε. κατά, αποχές, εγκρίνεται. Επόμενη έκθεση, Χιμπνερ. Μέσα επιμερισμού του κινδύνου για τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν ή απελούνται από σοφαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική του σταθερότητα. Ψηφίζουμε 17 τροπολογίες της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης μαζί και τις 17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Η τροπολογία υπαριθμών 24 τώρα με ονομαστική κλίση που αρχίζει. Πέρας. Απορρίπτεται η τροπολογία 24. Για να ψηφίζουμε την 25. Ψήφι... Ε, πάλι ονομαστική. Αρχίζει τώρα η ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται και αυτή η τροπολογία. Κύριε Καρόνα. Σενιόρα Καρόνα, καπηγείο παλάβρα. Ζητήσατε το λόγο. Σενιόρ Καρόνα. Ο κύριος ζητάει συγγνώμη, ο πρόεδρος. No. Α, sì, signor Speroni. Ο κύριος Σπερώνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι στις οθόνες έλεγε ότι αρχίζει η ψηφοφορία στις 12 και 10 ενώ ξεκινήσαμε από τις 12 και 09. Και να σας πω ότι και τα ρολόγια της αίθουσας είναι, πάνε μπροστά δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σπερώνη για την ε, χρονική σας ακρίβεια. Ψηφίσουμε τώρα την τροπολογία υπαριθμών 19. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 21. Με ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα για την τροπολογία 21. Πέρας. Και η τροπολογία απορρίψεται. Τροπολογία 14. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 22. Με ονομαστική κλίση. Αρχίζει τώρα. Απορρίπτεται. 16. Ψήφι ΠΕΡΑ κατά τροπολογίας αποχής συγκρίνεται. Η τροπολογία 23 με νομαστική κλίση που αρχίζει τώρα ψηφοφορία. Απορρίπτεται και αυτή η τροπολογία. πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική κλίση που αρχίζει τώρα. Εγκρίνεται. Και το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος με ονομαστική και πάλι κλίση αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Επόμενο σημείο. Πρόταση ψηφίσματος της Ενωτικής Αριστεράς και Βόρειας Πράσινης Αριστεράς για τη γνώμη του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη συμβατότητα με τις συνθήκες της Συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ της και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρήση και διαβίβαση φακέλων ονομάτων επιβατών. Ψηφίζουμε. Ψήφι υπέρ του ψηφίσματος αυτού κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε την έκθεση της κυρίας Σινετβέλτ για το ίδιο θέμα, το PNR. Ορίστε. Η συγκήτρια. Κυρία Νιτβέλτ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε απαντώντας σε μια σειρά συναδέλφων που ήταν σε σύγχυση για το τι ψηφίζουμε. Αν είστε υπέρ της συμφωνίας θα πρέπει να υπερψηφίσετε την έκθεση. Αν είστε κατά της συμφωνίας θα πρέπει να καταψηφίσετε την έκθεση. Θα ήθελα να βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως σύγχυση. Muchas Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, κύριε Νετβέλτ, ψηφίζουμε λοιπόν την πρόταση χωρίς τροπολογίες με ονομαστική ψηφοφορία που αρχίζει τώρα. Σε φιάβρα Πέρας. Εγκρίνεται με μεγάλη διαφορά. Pasamos al informe. Ναι, κύριε Ρασβέλτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για τα πρακτικά και για τη διοίκηση θα ήθελα να πω μόνο το εξή. Θέλω να αποστασιοποιηθώ από την έκθεση και να αφαιρέσω το όνομά μου γιατί είναι αντίθετο ε, το αποτέλεσμα προς τη σύσταση. Με ευχαριστώ. Ψηφίζουμε τώρα την της κυρία Στάισεν κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιριών. 37 τροπολογίες ψηφίζουμε της αρμόδιας επιτροπής. Ψήφι Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία παριθμών 41. Ψήφι Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 42. Τροπολογία ψυχή Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 43. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 39 με ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα ψηφοφορία. Πέρασε υπορρίψετε η τροπολογία αυτή. Ψηφίσουμε την τροπολογία υπαριθμών 14 τώρα. Ψηφιπέ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και καταπίπτει συνεπώς η 40. Το σύνολο της πρότασης όπως τροποποιήθηκε, Ψήφιπε. Κατά. Δεν είναι σαφές. Παρακαλώ, χρειάζεται επαλήθευση ηλεκτρονική για το σύνολο της πρότασης. Αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται, σαφώς. Και τώρα το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος με ονομαστική κλίση που αρχίζει τώρα. εγκρίνεται σαφώ και το ψήφισμα. Έκθεση Λούλινγκ. Για την κοινή ενοποιημένη, α, για τη φορολογία των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας. 42 τροπολογίες αρμόδιας επιτροπής. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 23 με ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να κάνουμε μια παλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 34. Υπέρ. Σηκώστε τα χέρια σας παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Είναι οριακή η ψηφοφορία να το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και αυτή. Και τώρα ψηφίζουμε την 40 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Και τώρα την 63 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Σαφέστατα. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Φοβάμαι ότι πρέπει να το επαληθεύσουμε και αυτό. Άρχεται η ψηφοφορία. Σε cierra votación. Πέρασε ψηφοφορία. Η ισοψηφία Επομένως, απορρίπτεται. Πενήντα δύο υπέρ. Συγγνώμη, η 52 είναι αυτή που μόλις ψηφίσαμε. Συγκινήθηκα από την ισοψηφία αυτή και καταλαβαίνετε. 53 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Σε Πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται, σαφέστατα. Και τώρα ψηφίζουμε την 55 υπέρ. Σηκώστε τα χέρια σας παρακαλώ υπέρ κατά αποχές να το επαληθεύσουμε άρχεται η ψηφοφορία Σε cierra votación. της ψηφοφορίας; Εγκρίνεται. Ψηφίσουμε τώρα Την τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Το μισό ημικύκλου δεν σήκωσε ούτε καν το χέρι του. Σας παρακαλώ, το επαληθεύουμε λοιπόν, να έρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 8. Πέρασε τη ψηφοφορία και η τροπολογία εγκρίνεται σαφέστατα. Και τώρα ψηφίζουμε την τροπολογία 51 υπέρ. Κατά. Άρχεται η ψηφοφορία για να το επαληθεύσουμε. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται με μεγάλη διαφορά. Ψηφίζουμε τώρα τη 16, όχι αυτή καταπίπτει. Περνάμε λοιπόν στο σύνολα της πρότασης ως τροποποιήθηκε υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται και Ψηφίζουμε και το νομοθετικό ψήφισμα με η ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην κυρία Λούλινγκ. Ωραία λοιπόν. Περνάμε στην πρόταση ψηφίσματος για την εξέβρεση συγκεκριμένων τρόπων καταπολέμησης φορολογικής απάτης Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται, σαφέστατα. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία υπαριθμών 3, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Την 7 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας εγκρίνεται με μεγάλη διαφορά. Τροπολογία 1 υπέρ. Σηκώστε τα χέρια σας παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 4 αποσύρθηκε και ψηφίζουμε την αιτιολογική σκέψη ε σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Το πρώτο τμήμα εγκρίνεται με μεγάλη διαφορά. Δεύτερο τμήμα τώρα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη F, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη G, με ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε τη ψηφοφορίας εγκρίνεται σαφέστατα. Και τώρα η πρόταση ψηφίσματος στο σύνολό της με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μεγάλη διαφορά. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα στις επεξηγήσεις ψήφου.